Let's Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ξανά τη συνεδρίαση. Βλέπω δύο συναδέλφους και εγώ είμαι ο τρίτος, τρία άτομα. So we have, uh, we now come Περνάμε τώρα στη συζήτηση για την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΑΦΕΤ για την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Οικονομικό Έτος 2018. Ως συνήθως προτείνω η συζήτηση να γίνει από ε, κοινού, να γίνει και για τα δύο θέματα. Σε ό,τι αφορά την ε, δημοσιονομική απαλλαγή στην Επιτροπή ΑΦΕΤ έχουμε επιφορτιστεί με το, την αρμοδιότητα να εξετάσουμε και να ασκήσουμε έλεγχο στο πώς δαπανώνται τα ε, ευρωπαϊκά κονδύλια. Ταυτόχρονα πρέπει να αποφύγουμε ε, τις υπεραπλουστεύσεις και να λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερη φύση της εξωτερικής δράσης. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που ο εισηγητής κ. Μεϊμαράκης έχει θετήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση και ε, έχει δώσει σημασία στα σημαντικά θέματα. Γι' αυτό λοιπόν θα του ε, ζητήσω να πάρει το λόγο και να μας παρουσιάσει την νομοδότηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και όσους ε, εργάστηκαν για τις νομοδοτήσεις, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την εξαιρετική έκθεσή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές και πολύπλευρες προκλήσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ σήμερα να είμαστε ενωμένοι, να πρωταγωνιστούμε στη διεθνή σκηνή, αναπτύσσοντας και ξεκάθαρες θέσεις στα κέρια ζητήματα που μας αφορούν. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να δοθεί βεβαίως η ευκαιρία και σε αντιπροσώπους μικρότερων χωρών να μπορούν να εξελιχθούν σε υπηρεσίες όπως η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και να προασπίσουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Είναι επίσης απολύτως απαραίτητο να ενισχύσουμε το έργο της υπηρεσίας ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στα αυξημένα πλέον καθήκοντα που έχει κληθεί να αναλάβει. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα πως στηρίζω απόλυτα τις εισηγήσει του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η αποκλειστική μας προτεραιότητα είναι η εκπροσώπηση των πολιτών. Είναι μέγιστη ευθύνη μας λοιπόν να διασφαλίσουμε στο σκέλος που μας αναλογεί ότι τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου πρέπει να χρησιμοποιούνται με διαφάνεια και να παράγουν αυτά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στι περιπτώσει όπου τα χρήματα αυτά προορίζονται για τι εργασίες μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός πως οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να προσκομίζουν στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο όλα τα έγγραφα που χρειάζονται προκειμένου να εκτελέσει υπεύθυνα και αποτελεσματικά το έργο του. Προσβλέπω λοιπόν σε μια αγώνιμη και επικοδομητική συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές, ώστε να καταλήξουμε σε ένα καλό και χρήσιμο αποτέλεσμα για την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Now if I'm... Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάζω γύρω μου και νομίζω πως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δει στο λόγο. Παρακαλώ. Αδελφοί, δεν θα ακρηγορήσω. Άλλο ο συνάδελφο έχει και μια πολύ καλή δουλειά και οι δύο γνωμοδοτήσει που μα παρουσίασε σήμερα έχουν τα βασικά σημεία που πρέπει να αναφερθούν στη διαδικασία απαλλαγή τη Επιτροπή για τη χρήση του 2018. Σε δύο μόνο σημεία θα ήθελα να σταθώ. Σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε γενικές γραμμές δεν εντοπίζονται προβλήματα διαφάνειας, με εξαίρεση όμως έργα που χρηματοδοτούνται μένα από εμάς, αλλά μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Ίσως εκεί θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει ξανά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και να υπάρξουν βελτιώσεις όπου είναι αναγκαίο. Επιπλέον, σχετικά με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ένωσης, θα ήθελα να σημειώσω πως συμφωνώ με τις διαπιστώσεις του εισηγητή και να τονίσω από την πλευρά μου την ανάγκη ενίσχυσης της υπηρεσίας με προσωπικό που δεν θα προέρχονται μόνο από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών, αλλά θα έχουν σταδιοδρομήσει και οι ίδιοι στα ευρωπαϊκά όργανα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για θέσεις ευθύνης και τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών σε τρίτες χώρες. Είμαι σίγουρος ότι χάρη στην πολύχρονη εμπειρία του συγητή μας που ξεκινάει από τη Βόλβη και φτάνει μέχρι τις Βρυξέλλες, θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Εφόσον λοιπόν ε, ακούσαμε όλα αυτά, τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχουν άλλοι σκιώδεις εισηγητές που θα ήθελαν το λόγο ή όσοι θέλουν να μιλήσουν εκ μέρους τους. Όχι, δεν βλέπω κανέναν. Θα θέλατε να απαντήσετε στη δήλωση του συναδέλφου ή να το αφήσουμε. Ωραία, εφόσον δεν έχουν ζητήσει άλλοι συνάδελφοι το λόγο, μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Η καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών είναι η 10η Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Το σημείο 18 είναι τα διάφορα. Θα ήθελε κάποιος να συζητήσουμε κάτι στα διάφορα. Όχι. Επόμενη συνεδρίαση στις 16 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Στρασβούργο και μετά το νέο έτος στις 20 Ιανουαρίου από τις 3 ως τις 6.30 και στις 21 το πρωί και το απόγευμα. Παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι τις τελευταίες ημέρες πως το Ιράν τα πράγματα είναι δραματικά. Η κατάσταση γίνεται όλο ένα και πιο βίαιη. Ίσως θα μπορούσαμε την επόμενη φορά να συζητήσουμε λίγο για το Ιράν και ίσως η υπηρεσία θα μπορούσε να μας δώσει πρόσθετες πληροφορίες. Από όσο γνωρίζω, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 750 νεκρούς, πάνω από 12.000 τραυματίες και συλληφθέντες. Ναι, από όσο γνωρίζω και εγώ, τα νούμερα αυτά δυστυχώς ε, ισχύουν. Το καθεστώς γίνεται ολιώνα και πιο κατασταλτικό. Υπάρχουν μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα και θα μεταφέρω το έτοιμά στη γραμματεία για, και στο Προεδρείο για να δούμε ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για να το συζητήσουμε. Μικρόφωνο ανοίξτε παρακαλώ. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε την κατάσταση στο Ιράν όχι μόνο εξαιτία των εξελίξεων, αλλά και σε ένα γενικότερο πλαίσιο για την περιοχή αυτή, διότι υπάρχει και η περίπτωση της ε, Ιεμένης, της Συρίας, του Λιβάνου, βρίσκονται ε, όλες αυτές οι περιοχές εκεί κοντά και τα πράγματα είναι πολύπλοκα, αλλά παρακαλώ να συζητηθεί το θέμα του Ιράν. Ωραία, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο, νομίζω πως μπορούμε να λήξουμε τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς. Λίγη συνεδρίαση.